περνούσε κατά πολύ το ύψος των υπολείπων και θα θέλαμε να στείλουμε συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Ε, Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Έχω πάρει από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών μία αίτηση για ορισμούς σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κατάλογος των διορισμών αυτών θα προσαρτηθεί στα πρακτικά μας. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί αυτοί οι διορισμοί όταν γίνει η έγκριση των πρακτικών. Επίσης βάσει του άρθρου 3 και της παράγραφης 3 και 4 του άρθρου 3 η Νομική Επιτροπή συνεδρίαση της 20 και 26 Ιανουαρίου 2011 έλεξαν την εντολή της Μαρία Ιριγκοϊέν Πέρεθ, του κυρίου Φιλίπ Μπουγιάν και της κυρίας Αγνές Λεμπράν. Ομόφωνα προέτεινε να θεωρηθεί ότι έχει ελεγχθεί η εντολή της κυρίας των τριών αυτών ατόμων, να θεωρηθεί ότι είναι έγκυρη η εντολή τους. Τη κυρία Σιριγόιεν Πέρε από 16 Νοεμβρίου 2010, του κυρίου Φίλιπ Μπουγιάρ από τι 15 Δεκεμβρίου και τη κυρια αγνε Αγνές Λεμπρέν από 1η Ιανουαρίου 2011. Προτείνω λοιπόν να θεωρήσουμε ότι, έχουν, ότι είναι έγκυρες οι εντολές αυτών των τριών βουλευτών. Έχετε σχόλια. Εάν όχι, ούτως απεφασίστη. Επίση, βάσει το άρθρο 216 του κανονισμού, η αρμόδια επιτροπή έχει υποβάλει δύο ορθωτικά σε σχέση με ένα κείμενο που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2010 εν ώψη της έγκρισης του κανονισμού για την ε, πρωτοβουλία πολιτών Έχει γίνει μια τροποποίηση λοιπόν αυτή τη ε, θέση βάσει του άρθρου 216 παράγραφο 4 του κανονισμού. Αν στι επόμενε 48 ώρε οι πολιτικέ ομάδε, οι 40 βουλευτέ δεν ζητήσουν να ψηφιστεί αυτή η τροποποίηση, το διορθωτικό αυτό θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί. Βρίσκεται στους φακέλους σας <clears throat> και επίση και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Πρόκειται λοιπόν για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το έγγραφο που εγκρίναμε στις 15 Δεκεμβρίου 2010 σε πρώτη ανάγνωση. Έχουμε τώρα τροποποιήσει στην ημέρησια διάταξη. Το τελικό σχέδιο της ημέρησιας διάταξης ενεκρίθη από την συνέλευση των Προέδρων Βάση του άρθρου 216 και με τη συμφωνία των πολιτικών ομάδων. Θέλω να σας πληροφορήσω για αυτές τις αλλαγές μονάχα και θα αναγνώσω τις προτάσεις αυτές που έχουν διατυπωθεί. Είναι πέντε προτάσεις. Έτυχαν συμφωνίες από τις πολιτικές ομάδες και τις διαβάζω για την έγκριση της Ολομέλειας. Πρώτον, ε, ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα κάνω μια δήλωση για την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της γενοκτονίας των Ρωμά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και θα ακολουθήσει δήλωση του Συμβουλίου από την Κομισιόν και θα λάβουν το λόγο εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων για το ίδιο θέμα αυτό, δηλαδή για τη γενοκτονία των Ρωμά στον Δεύτερο Παγκοσμίου Πόλεμο. Δεύτερον, για σήμερα. Η επικεφαλίδα της συζήτησης για την κατάσταση στην Τινησία τροποποιήθηκε και έχει ως εξή. <clears throat> Δήλωση της Αντιπροέδρου της Κομισιόν και υπά της εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικά Θέματα και Πολιτική Ασφάλειας επί της καταστάσεως στη Μεσόγειο, ιδιαίτερο στην Τινησία και στην Αίγυπτο. Τρίτον, η τρίτη αλλαγή για σήμερα. Η ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τα ψηφίσματα που αφορούν την Τινησία θα γίνει αύριο όπως έχει ήδη προγραμματιστεί. Η ψήφιση όμως ψηφισμάτων σε σχέση με την ΑΕΤΟ θα γίνουν στη δεύτερη σύνοδο Ολομέλειας του Φεβρουαρίου, δηλαδή στο Στρασβούργο. Τέταρτη πρόταση αλλαγής. Η συζήτηση σε σχέση με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την άνοδο της τιμής των τροφίμων αναβάλλεται για τη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα αντικατασταθεί από δηλώσει του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τον διορισμό υψηλών αξιωματούχων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών που θα ακολουθηθεί και από ομιλίες των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Με σύντομη συζήτηση λοιπόν για το θέμα αυτό του διορισμού υψηλών αξιωματούχων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τα οικονομικά θέματα. Την Πέμπτη επίσης η έκθεση Σπερώνη για την αίτηση άρσεως της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Ταμάς Ντόιτς θα συμπεριληφθεί στον χρόνο ε, ψηφοφοριών. Θα ψηφιστεί δηλαδή περίπου αύριο το μεσημέρι στις 12. Έχετε κάποια σχόλια σε, σχέση με αυτές τις τροποποίησεις. Όχι. Τότε, βάσει τις συμφωνίες που επιτέχει μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αυτές οι αλλαγές στην ημέρηση διάταξη έχουν εγκριθεί. Έχετε το λόγο. Διαδικαστικό θέμα. Γιάν Πάσκου. Διαδικαστική παρέμβαση. Θα ήθελα να ζητήσω να προταχθούν οι ομιλίε ενό λεπτού, γιατί στις τελευταίες συνόδους Ολομέλειας έχουν ε, τεθεί στο τέλος του χρόνου της Ολομέλειας και όλο και λιγότερα άτομα συμμετέχουν στο χρόνο των ομιλιών ενός λεπτού και λυπάμαι για το γεγονός αυτό. Ίσως λοιπόν πρέπει να εξετάσετε να προταχθούν οι ομιλίες του ενός λεπτού για να μπορούμε να συμμετέχουμε πιο πολυπληθείς σε αυτές τις συζητήσεις όπως κάναμε και νωρίτερα. καταγράφουμε αυτό το οποίο λέτε. Ξέρω ότι θα γίνει και μια συζήτηση για το θέμα αυτό και θα ληφθούν οι αρμόδιες αποφάσεις από την συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει μεταξύ των πρόεδρων των πολιτικών